Dear colleagues, good afternoon. Please Καλησπέρα συνάδελφοι, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε συνεδρίασή μας. Ετοιμάστε τα ακουστικά σας, διότι θα περάσω τα λιφωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας πω ότι είμαι η κυρία Πλίνκεβιτσιούτα και έχω την τιμή ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής να επιτελέσω τα καθήκοντα της προσωρινής Προέδρου. Καθήκον μα λοιπόν σήμερα είναι να εξελέξουμε τα μέλη του Προεδρείου, τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους. Τέσσερις στον αριθμό, Αντιπρόεδρε. Βάσει του άρθρου 213 του κανονισμού. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω τα ονόματα των ε, αναπληρωτών Κόπατς, Λόκατς, την κυρία Ροφκατσεύσκα, την κυρία Πιετικά να αντικαθιστούν επίση. και η κυρία Έντπεργκερ Ποπάνα, τον κύριο Ούρτασουν. Και τώρα να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία για την εκλογή του Πρόεδρου. Έχουμε απαρτία. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ψηφοφορία και τώρα να ακούσουμε τους υποψηφίου. Το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την ομάδα των Συλληστών και Δημοκρατών προτείνουμε τον υποψηφιό μας την Εύενη Ρέγνερ από την Αυστρία. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, λέει ο Πρόεδρος, να ρωτήσω την κυρία Εύελιν Ρέικνερ κατά πόσον είναι σύμφωνη με την υποβολή της υποψηφιότητάς της. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Στη συνέχεια, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η κυρία Ρέγνερ είναι τακτικό μέλλον, έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων, καθώς και την ε, σχετική δήλωση για την καλή συμπεριφορά. Και μιας και δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος για τη θέση της Πρόεδρου, θα πρότεινα διαβοήσει να ψηφίσουμε την κυρία Ρέγνερ.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 So, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Πριν πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στις υποψηφιότητες για τις θέσεις των αντιπροέδρων, θα ήθελα να κάνω μία μικρή εισαγωγή για μένα και τις προθέσεις μου. Εύλιν Ρέγνερ λέγομαι, είμαι Αυστριακή, είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και 10 χρόνια. Έχω δηλαδή πολλή εμπειρία και κρατώ αμύωτο το ζήλο μου για το ευρωπαϊκό μας έργο. Είμαι φεμινίστρια, είμαι συνδικαλίστρια, έχω δύο παιδιά. Ξέρω λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο για όλους εδώ εμάς αυτή την αίθουσα. Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό ε, και θα το κάνουμε στην Επιτροπή Γυναικών μαζί σας. Θέλω να πολεμήσω για την Ευρώπη που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Μια Ευρώπη όπου οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν παρενόχληση, μια φεμινιστική Ευρώπη και δεν θέλουν να υπάρχουν διαφορές στο, ποιος στο ποιον θα αγαπούμε. Θέλω να σταματήσουμε τις διακρίσεις απέναντι στους ΛΟΑΤ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ως πρόεδρος. Και με μεγάλη τιμή θα προεδρεύσω σε αυτή την Επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι η Επιτροπή Γυναικών είναι ένα σωστό χώρο για να συνεχίσουμε το σημαντικό αγώνα για την ισότητα. Καταρχά, και σημαντικό, οικονομικά πρέπει να είμαστε ανεξάρτητε. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Όποιο κι αν είσαι, άντρα, γυναίκα, όποιον και να αγαπά, θα πρέπει να το πετύχουμε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε χάσμα στο μισθό ανδρών και γυναικών. Και κάτι άλλο. Αυτό είναι τμήμα του DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε. Θα πρέπει να πολεμήσουμε την αντίδραση απέναντι στις γυναίκες και στους ΛΟΑΔ και τα δικαιώματά τους εδώ στην Ευρώπη. Είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και είναι η ευθύνη μας, ούτως ώστε οι γυναίκες παντού σε όλη την Ευρώπη να κάνουν τις δικές τους επιλογές πάνω στα σώματά τους. Πρέπει να πολεμήσουμε για να πετύχουμε ισότητα των φύλων στην οικονομική, στην οικονομική σφαίρα και στην πολιτική σφαίρα και στις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις. Ως ε, εισηγήτρια για τις γυναίκες στα Δουσού περιμένω εδώ και έξι χρόνια, πολύ καιρό, να σταματήσει το Συμβούλιο το μπλοκάρισμα πάνω σε αυτό το θέμα για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Αλλά εμείς θα το καταφέρουμε γιατί δεν θα σταματήσουμε. Όλοι μαζί, όπως είμαστε και τώρα, το διεκδικούμε, το θέλουμε. Χρειάζομαι την υποστήριξη όλων σας και την υποστήριξη βεβαίως των αντιπροέδρων που θα εκλέξουμε πάρα αυτά. Πάμε λοιπόν μετά τα αυτά στο επόμενο βήμα της ημερήσιας διάταξης, την εκλογή των αντιπροέδρων. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό, να μην ξεχάσουμε τίποτα, με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να έχουμε την ε, απαιτούμενη απαρτία. Υπόθηκε ότι την έχουμε. Και τώρα, θέλουμε να εκλέξουμε τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αντιπρόεδρο και να δούμε ποιε είναι οι κατάλληλε υποψηφιότητε. Λοιπόν, ποιο θα προτείνει του υποψήφιου για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Από την QNGL, Γιωζένια Ροντρίγκε Πάλοπ είναι ε, η υποψήφια. Εουχένια Rodríguez Πάλοπ. Συγγνώμη. Κυρία Ροδρίγκεθ Πάλοπ, επιβεβαιώνετε ότι δέχεστε αυτή την υποψηφιότητα. Βεβαίως, ευχαριστώ. Είσαστε πλήρες μέλος, τακτικό μέλος δηλαδή της Επιτροπής Γυναικών. Έχετε υπογράψει τον κώδικα διοντολογίας και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων Θα ήθελα λοιπόν να σας εκλέξουμε διαβοής. Παρακαλώ, όσοι είναι υπέρ της υποψήφιας, να χειροκροτήσουν. Συγχαρητήρια. Μπορείτε να έρθετε εδώ στο Προεδρείο. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, στην επόμενη εκλογή. Um, Συγχαρητήρια. Περνάμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου. Ποιος θα προτείνει τους υποψήφιους, παρακαλώ. Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά προτείνω την κυρία Γκουεντελίν Δέρβες Κόμφιλτ για, τη δεύτερη θέση, για το δεύτερο, την θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Κυρία Δελμπός ε, Κόρφιλντ. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Ναι, είσαστε τακτικό μέλος της Επιτροπής. Έχετε υπογράψει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τον κώδικα συμπεριφοράς. Θα ήθελα επίσης να σε εκλέξουμε διαβοής, όπως και πριν. Όπως κάναμε και πριν. Η του πρώτου αντιπρόεδρου, δηλαδή. So, congratulations and, uh... Συγχαρητήρια, καλώς ήρθατε και εσείς εδώ στο Προεδρείο μεταξύ των Αντιπροέδρων. Committee in Επόμενη θέση. Θα εκλέξουμε τον τρίτο αντιπρόεδρο. Η γνωστή διαδικασία. Ποιο θα προτείνει τον, τρίτο, τον υποψήφιο για, τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Εκ μέρου του ΕΛΚ, Elizabeth η κυρία Ελίζαμπεθ Βόζενμπεργκ, για τη θέση αυτή. Κυρία Βόζεμπεργκ, συμφωνείτε? Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Δέχομαι την υποψηφιότητα. Είσαστε τακτικό μέλος της Επιτροπής. Υπογράψατε τον κώδικα διοντολογίας και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Προτείνω να κάνουμε όπως και πριν, να σας εκλέξουμε διαβοής. Ελάτε και εσείς στο Προεδρείο. We one vice president is missing. Και μας λείπει ένας αντιπρόεδρος. Βλέπετε πολλές γυναίκες στο Προεδρείο. Υπάρχει μια άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του τάρτου αντιπροέδρου. Ναι. Νομίζω ότι είναι, ίγκη και ώρα για να εκλέξουμε και έναν άντρα. Από την ομάδα των σοσιαλιστών προτείνω το Ρόμπερτ Πίρντον από την Πολωνία. Ρόμπερτ, συμφωνείς με την πρόταση? Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλες τις συναδέλφους. που εξελέγησαν. Είμαι ο τελευταίος. Και επειδή είμαι ο τελευταίος και μοναδικός, αισθάνομαι συνήθως όπως αισθάνονται οι γυναίκες. Βεβαίω, δέχομαι την υποψηφιότητα, με χαρά και τιμή. Σύμφωνα λοιπόν ε, με τον κανονισμό, μπορώ να επικυρώσω ότι έχει υπογράψει το κώδικα διοντολογία αλλά και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων ότι είσαι τακτικό μέλος της Επιτροπής και ότι μάλιστα υπάρχει στη σύσταση της, του Προεδρείου η πολυμορφία που ζητάει το Κοινοβούλιο και τώρα νομίζω θα ήθελα επισήμω να σε εκλέξουμε διαβοής πλέον είσαι ο τέταρτος αντιπρόεδρος. Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Θα ήθελα να πω ότι ε, χαίρομαι που, ε, για, τη, για τη σύσταση ε, του Προεδρείου και τη σύσταση της Επιτροπής. Θα είμαστε πολύ ισχυροί για να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας και μάλιστα ανυπομονώ ανυπομονώ να κάνω όλα αυτά που, έχουμε αποφασί... που, που, προβλέπονται με, με μαζί σας. Κάποιες ανακοινώσεις που θα ήθελα να σας πω. Αφενός, η επόμενη συνεδρίαση α, έχετε λάβει μάλιστα μέσω email ε, τις προσεχείς συναντήσεις μας της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε θετείτε ε, το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει. Αν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αν όχι, τότε ε, υιοθετείτε. Το επόμενο ε, ζήτημα είναι το γλωσσικό προφίλ. Επίσης έχετε λάβει μέσω email το, το γλωσσικό προφίλ της, ε, ε, της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις τότε επικυρώνεται και αυτό. Τέλος, σας μοιράστηκε ένα αρχείο ως καλωσόρισμα. Επίσης ε, μπορείτε να το βρείτε και αυτό στο διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες. Η προσεχής ε, συνάντηση, η προσεχή συνεδρίαση θα είναι στις 24 Ιουλίου στις 9 στις Βρυξέλλες. Ε, υπάρχει ακόμα μια συνεδρίαση. Ελπίζω ότι θα είστε στην επόμενη συνεδρίαση πριν φύγετε για διακοπές. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με αυτά τα λόγια την συνεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ, ας δουλέψουμε όλοι μαζί.